Good afternoon everybody. Καλησπέρα σας. I could use my hammer. Έχω και σφυράκι, αλλά δεν νομίζω θα μου χρειαστεί, να μου χρειαστεί. Καλώς ορίσατε. Ελπίζω όλοι να περάσατε καταπληκτικές διακοπές. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μάλιστα, εγκρίνθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσεις. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ε, μεταδίδεται από το διαδίκτυο απευθεία στη συνεδρίασή μας για τις ακροάσεις των επιτρόπων, ε, πιο πρόσφατα στοιχεία που έχω υπόψη μου είναι ότι μου είπαν ότι την Τετάρτη το βράδυ να μην κανονίσω τίποτα γιατί θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Οπότε μάλλον θα ακούσουμε νέα για, το, για πρόσωπα, ονόματα και χαρτοφυλάκια ε, από μέχρι την Τετάρτη, νωρίς την Τετάρτη. Και η έκτακτη αυτή ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συγκαλείται για να αποφευθούν οποιασδήποτε παρεξηγήσεις τώρα και συγκρούσεις περί αρμοδιοτήτων. Έχουμε Έχουμε λάβει και επιστολές. και προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αποσταλεί για να παραμείνει στην, Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικά η ε, προστασία των καταναλωτών να συνεχίσει να δίδεται ιδέουσα προσοχή και να δούμε και πώς η δική μας Επιτροπή που ασχολείται με την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών ε, πώς επαναπροσδιορίζεται ας πούμε ως προς τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες με την νέα εντολή και την νέα θητεία. Έχουμε συνεργασία και με την Επιτροπή Οικονομικών και με την Επιτροπή Βιομηχανίας σε διάφορα θέματα αλλά και σε θέματα ε, εσωτερικού εμπορίου, έτσι. Ωραία. Αυτά για να σας ενημερώσω. Μόλις μάθω τίποτα νεότερο για τις ημερομηνίε, ε, τις ε, πιθανές των ακροάσεων, θα σας ενημερώσουμε. Γνωρίζω ότι στο παρελθόν τα μέλη της Επιτροπής μας συμμετείχαν σε πάρα πολλές ακροάσεις και είχε ασκηθεί και τεράστια πίεση χρονική για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτές τις ακροάσεις. Παρακαλώ όμως προσπαθήστε να συμμετέχετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, ως αρμοδιότητα και ευθύνη του Κοινοβουλίου. Και πριν από πέντε χρόνια είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πολλές ακροάσεις και το επιδίωξα για να βολιδοσκοπήσω τους ε, διαφόρους υποψηφίους και να τους αξιολογήσω και είχα και μια καλύτερη εικόνα γενικότερα. Ah, για τις ε, ηλεκτρονικές συνεδριάσεις σας θυμίζω ότι είμαστε επιτροπή χωρίς έγγραφα και μπορείτε να μπείτε από την εφαρμογή αυτή της ηλεκτρονικής επιτροπής e-meeting για να έχετε όλα τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Τα γνωρίζετε όλα αυτά εξάλλου. Και θα ήταν ενδεχομένω χρήσιμο να εκπαιδεύσουμε και τους βοηθούς ε, σε αυτό το θέμα. Ωραία. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης ή των προηγούμενων συνεδριάσεων. Ερωτήσεις. Γκρίνονται. Ωραία. Και μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσω τότε στις ψηφοφορίες. The first vote is on delegation of powers to the coordinators. Κατ' αρμοδιότητες συντονιστές στη συγκεκριμένη mm. περίπτωση σύμφωνα με το 205 2. Δίνεται η δυνατότητα στον Πρόεδρο να συγκαλεί συνεδριάσεις των συντονιστών και οι συντονιστές να παίρνουν αποφάσεις εξ ονόματος της Επιτροπής σε σχέση με κατανομής εκθέσεων και ορισμό εισηγητών. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επιλέξει να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες εφόσον το επιθυμεί στους συντονιστές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία απαιτείται. Παρακαλώ πάρτε τις κάρτες σας. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. ένας δεν έχουν ακόμα ψηφίσει. Τρεις ακόμα. Or Τέλος. 25 υπέρ λοιπόν. Τρεις κατά, δεκτή. Περνάμε τώρα στην έγκριση του γλωσσικού προφίλ. Να πω εδώ ότι η πρόθεσή μας είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αίθουσα για να καλύψουμε όλες τις γλωσσικές ανάγκες και των 22 διαθεσίμων δηλαδή γλωσσών. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Ρώτησα από τη Γραμματεία να ελέγξει για μια ακόμη φορά ότι χρειαζόμαστε και τις 22 γλώσσες, ότι έχουμε μέλη δηλαδή για τις γλώσσες αυτές. Αυτό θα είναι χρήσιμο. εάν τυχόν βρούμε ότι η διερμηνία παρέχεται για μέλη τα οποία δεν είναι παρόντα τακτικά, τότε ίσως θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Θα πρέπει να μας δηλώνουν αν δεν σκοπεύουν να είναι παρόντες και να μας ενημερώνουν, να ενημερώνουν τη γραμματεία, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούμε αδίκως τους διευμηνείς. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της παρουσίας της διευμηνίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο κόσμος να ακούει άμεσα και να κατανοεί αυτά τα οποία λέμε. Έχετε το λόγο. Η κυρία Γιά Κονσάρη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτά που είπατε, η τεκμηρίωση την οποία παρουσιάσατε είναι ο λίγων ιδιόρυθμη. Είπατε ότι η παροχή ε, διερμηνίας οφείλεται ή εξαρτάται μάλλον από το μέγεθος της αίθουσας. Ε, δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Ε, μπορεί κάποια περίπλοκα θέματα να τα συζητάμε σε μικρές αίθουσες και κάποια απλούστερα σε μεγάλες αίθουσες. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι οι αρχές τις οποίες εσείς καταθέσατε ε, πράγματι πρέπει να υπάρξει εξοικονόμηση αλλά το να, θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να μην μεταφέρεται η συνεδρία σε μικρή αίθουσα και έτσι να μην υπάρχει και διευμηνία. Κοιτάξτε, εγώ είπα ότι όλες θα ζητήσω όλες οι συνεδριάσεις να γίνονται σε αίθουσες με δυνατότητα 22 θαλάμων διερμηνίας για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Αλλά θα ελέγξουμε αν έχουμε ανάγκη όλες τις γλώσσες. Το θέμα είναι ότι αν όλες οι επιτροπές ζητούν ταυτόχρονα τη χρήση μεγάλων αιθουσών, τότε έχουμε κάποια προβλήματα. Θα το ζητήσουμε λοιπόν, θα το ελέγξουμε και ελπίζω να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και υποστηρίζω την ανάγκη σας σαν δραστήριο μέλλον, μέλος <laughs> συγγνώμη, της Επιτροπής μας να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας στην γλώσσα σας. Είναι σημαντικό επίσης και για τους καταναλωτές να παρακολουθούν από πρώτο χέρι τις συνεδριάσεις. Θέλω να προσθέσω ένα επιχείρημα σχετικά με τις γλώσσες, διότι μη λησμονείτε ότι δεν είναι μόνο τα μέλη που είναι παρόντα εδώ, είναι και οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις από το διαδίκτυο. Θα πρέπει να φροντίζουμε λοιπόν να διερμηνεύονται οι συνεδριάσεις σε όλες τις γλώσσες, ώστε και οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν το ότι συζητείται. εδώ. Μιλούμε κάθε φορά για την ανάγκη εγκύτητας στον πολίτη και ξαφνικά αρχίζουμε πάλι να βάζουμε εμπόδια ακριβώς εκεί, όπου τίθεται θέμα επικοινωνίας με τον πολίτη ή την πολίτη. Εκεί πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. This is not about cuts and savings, about whether or not... Δεν μιλώ για περικοπές, αλλά για εάν πραγματικά τη συγκεκριμένη γλώσσα τη χρησιμοποιούν τα μέλη. Καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλετε εσείς είναι να εξασφαλίσετε ότι θα μεταφράζετε στις 22 γλώσσες, έστω και αν δεν χρησιμοποιείτε μέσα στη συνεδρίαση μια γλώσσα. Αυτό βέβαια είναι διαφορετικό θέμα. Θα εξετάσω πάντως πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όπως είπα στην αρχή, θα ζητούμε πάντο, πάντοτε για λογαριασμό της Επιτροπής μας να έχουμε στη διάθεσή μας μεγαλύτερες αίθουσες με τη δυνατότητα μεταφράσεως 22 γλωσσών. Η κυρία Μεζόλα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα προκατακτικά που είπατε. Ένα χρόνο τώρα είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βλέπω αλλαγές και εξέλιξη. Βλέπω σε ορισμένες συνεδριάσεις να προστίθεται η μαλτέζικη γλώσσα και σε άλλες να αφαιρείται. Η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών ωστόσο είναι σημαντική για τους Μαλτέζους καταναλωτές. Έχουμε δύο από τους συνολικά έξι ευρωβουλευτές μας στην παρούσα Επιτροπή για την επόμενη πενταετία. Πολλοί πολίτες της χώρας μου παρακολουθούν τις συζητήσεις της Επιτροπής μας μέσα από το web stream. Και επαναλαμβάνω ότι το 1 τρίτο των ευρωβουλευτών μας, των Μαλτέζων ευρωβουλευτών μας δηλαδή, είναι παρόντες εδώ. Αυτό διότι μας παρακολουθούν οι Μαλτέζοι πολίτες. Thank you. And I know that Malta is on... Ναι, υπάρχουν ναι, και η γλώσσα της Μάλτας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 20 γλωσσών και στον κατάλογο των 18 γλωσσών. Κοιτάξτε, μας έχουν επιβεβαιώσει μεγάλες αίθουσες για την επόμενη συνεδρίαση για τον Οκτώβριο, για τις 5 και 6 Νοεμβρίου, για την συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου και της 3 ε, η και 4 η Δεκεμβρίου, προβλέπεται να γίνονται σε ε, αίθουσες με 20 θαλάμους και όχι 22. Θα δούμε τι θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αλλά προσπαθούμε πάντως. Θα σας ενημερώσω όσο μπορώ περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο γλώσσες οι οποίες θα εκπέσουν θα είναι τα λετονικά και τα εσθονικά. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε παρακαλώ τώρα στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου σημείου με τις προϋποθέσεις τις οποίες εκφράσαμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την έγκριση του γλωσσικού προφίλ της Επιτροπής μας, ηλεκτρονικά παρακαλώ. One more. Done. So that Λοιπόν, δεκτή. Τώρα, έγκριση των συστάσεων των ε, συντονιστών για τις εκκρεμότητα υποθέσεις. Αφορά 7 διαφορετικά θέματα όπου είχαν υιοθετηθεί ε, αποφάσεις σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης από το προηγούμενο κοινοβούλιο κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε με τις διαπραγματεύσεις ε, σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου. Έχω την έγκρισή σας παρακαλώ να προχωρήσουμε όπως ακριβώς το συστήνουν οι συντονιστές. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Sorry. Sorry, sorry. That's carried. Δεκτή η πρόταση. 28 υπέρ και 2 αποχές. Now, we move on to the vote on the budget. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η δημοσιονομική διαδικασία ήταν κάπως άτακτη λόγω των εκλογών που μεσολάβησαν. Απαιτήθηκε τεράστια προσπάθεια από την εισηγήτρια και τους σκιώδεις υπήρξαν μικρότερες προθεσμίες από ό,τι συνήθως Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει στο μέλλον να επανεξεταστεί, διότι πράγματι δεν είναι κάτι το οποίο δίνει τον απαιτούμενο χρόνο για συζήτηση για τα θέματα του προϋπολογισμού. Τα συζήτησα με την εισηγήτρια, συμφωνεί ότι δεν είναι ιδανική η διαδικασία λόγω των εκλογών, λόγω των χρονοδιαγραμμάτων για την έγκριση του προϋπολογισμού αναγκαστήκαμε να την ακολουθήσουμε. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος που έχει αναφερθεί σε αυτά, έχει εργαστεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις οι οποίοι έκαναν τεράστια προσπάθεια. Εμένα μου δώσαν δύο εβδομάδες για να εξετάσω την πρόταση λόγω ακριβώς του εκλογικού χρονοδιαγράμματος. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε και το πετύχαμε σε κάποια θέματα. Αυτό ήταν θετικό. Σε κάποιες άλλες τροπολογίες δεν μπορέσαμε να τις συμφωνήσουμε με αυτές και να τις υποστηρίξουμε αλλά έχετε απολύτως δίκιο ότι τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, το επόμενο έτος. Επίσης τίθεται εδώ το θέμα των λεγόμενων πιλωτικών προγραμμάτων. Αυτά τα οποία προκρίνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό αφορούν την ψηφιακή ατζέντα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ σημαντικούς τομείς στον τομέα των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αλλά η επόμενη γραμμή στον επόμενο προϋπολογισμό για τα πιλωτικά προγράμματα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και θα πρέπει να διαμορφώσουμε μία πρόταση επικοδομητική και συμβατή με τις προτάσεις των απαιτήσεων της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Και έτσι θα μπορέσουν να γίνουν δεκτές από αυτήν. Λοιπόν, ε, αυτά για το μέλλον, για το πώς μπορούμε συλλογικά να προωθήσουμε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία να γίνουν δεκτά συνολικά από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ όσους πήραν μέρος στην επεξεργασία των προτάσεων. Περιμένω την συζήτηση και την ψηφοφορία όταν γίνουν. Η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λέει η κυρία Γκραπίνη. Όπως είπε και η Κάθριν, δεν είχαμε χρόνο στη διάθεσή μας και εδώ τίθεται ένα θέμα αρχής, αν θέλετε. Εγώ έχω εργαστεί για τα θέματα των προϋπολογισμών ε, και στο παρελθόν ήμουνα και υπουργό προϋπολογισμού και θα πρέπει τον επόμενο χρόνο τα πράγματα να γίνουν με διαφορετικό παρακαλώ τρόπο θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες τις οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες της χώρες μας, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να επιληθούν οι ακρεμότητες, να ξεπεραστούν οι προβλεπόμενες δυσκολίες. Αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν φέτος στον ενεστώτα προϋπολογισμό, αλλά θα θέλαμε όμως η συζήτηση τον επόμενο χρόνο να είναι ε, επί της ουσίας ε, εφόσον δεν εργάζονται σωστά τα πιλωτικά προγράμματα θα πρέπει να σταθούμε καινοτόμα απέναντί τους και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχουν οι μικρομεσαίες κυρίως σε σχέση με την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, με την πρόσβαση σε δημόσιες προμήθειες κτλ. Πρέπει να συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα τα οποία θα λύσουν τα προβλήματα. Απτά. Καλώς λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Καταρχάς έχουμε μια ομαδική ψηφοφορία έτσι όπως συμφωνήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου από τις πολιτικές ομάδες. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν του πακέτου αυτού. Δέκα δεν έχουν ψηφίσει. Παρακαλώ το κόμμα των συντηρητικών τι κάνει εδώ, ναι ή όχι, δεν βλέπω το συντονιστή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Τέλος της ψηφοφορίας. 30 υπέρ της προτάσεως, 4 κατά της προτάσεως. Περνάμε τώρα στην ίδια την έκθεση. Υπάρχει από την εισηγήτρια μια προφορική τροπολογία. Κάθριν. Όλοι συμφωνείτε με την προφορική παρακαλώ διανατάσεως των χειρών. Δεκτή. Τώρα η τροπολογία 1. Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας κατέπεσε καθώς πέρασε η προφορική και θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την υπόλοιπη τροπολογία. Ψήφι πέρ. Against. Κατά. Απερίφθη. Η τροπολογία 2 έχει αποσυρθεί. Η 3 λοιπόν υπέρ. Κατά. Η 4 υπέρ, κατά, οι 5 υπέρ, συγγνώμη, εγκρίνεται λέει η πρόεδρος, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δηλαδή 3, 4, 5 εγκρίθηκαν και η τελική ψηφοφορία για το σχέδιο όπως τροποποιήθηκε Άλλοι πέντε παρακαλώ να ψηφίσουν. Let's close the vote. 28 for, for again. 28 υπέρ, 4 ε, ε, κατά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Um, just announcements on... Κάποιες ανακοινώσεις τώρα για τις επόμενες συνεδριάσεις μόνο. The next meetings of the committee will οι προσεχή συνεδριάσεις 24 Σεπτεμβρίου μέρα Τετάρτη, 9 το πρωί και 3 το απόγευμα και στις 25 Σεπτεμβρίου μέρα Πέμπτη συνεδριάζουμε στις 9 και ε, είναι πιθανό να έχουμε και κάποιες ψηφοφορίες εκεί. Είχε προγραμματιστεί και μια απογευματινή συνεδρίαση που μάλλον δεν θα χρειαστεί, θα τελειώσει το πρωί. Εντάξει, για να μπορέσετε να κανονίσετε τα ταξίδια σας και τις πτήσεις και για τις ακροάσεις θα σας πω το συντομότερο για τους ε, υποψηφίους επιτρόπους. Ευχαριστώ. Και τώρα συνεχίζουμε και κλεισμένων των θυρών χωρίς ε, δημοσιογράφους. Ε, βέβαια ε, το προσωπικό και η βοηθοί παραμένουν. Με την κυρία Φρανσουάζ Λεμπάη, ε, ε, Γενική Διευθύντρια ε, Εξωτερικών Σχέσεων.